Okay, colleagues, Μάλιστα, συνάδελφοι. Ας αρχίσει η συνεδρίαση. Καταρχάς, έχουμε την υιοθέτηση του σχεδίου της ημερίας διάταξης. Είναι όλοι σύμφωνοι. Μάλιστα. Έπειτα, η έκριση των πρακτικών της συνεδρίασης Τη 9 η και 10 η Ιουλίου 2012. Υπάρχουν ερωτήσεις ή αντιρρήσεις σε αυτό. Εάν όχι, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο, η σύναψη δημόσιων συμβάσεων, γνωμοδότηση από την κυρία Λίχτενμπέργκερ. Εύα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αρχίζουμε να ασχολούμαστε με έναν πολύ ενδιαφέρον τα φάκελο, οι δημόσιες συμβάσεις και τα κριτήρια ανάθεσής τους, δηλαδή ο καινούριος κανονισμός των, ε, της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε τον προσεχή χρόνο. Προσπάθησα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τροπολογίες μου και την αιτιολόγηση, και την και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους. Ε, προσπάθησα να συζητήσω και με τις υπόλοιπες επιτροπές της επί και να δω τι σχεδίαζαν εκείνες οι επιτροπές. Όσον αφορά τις αρχές, Η πρότασή μου είχε ως εξής. Εμείς να προσπαθήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κριτήρια για την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα των μεταφορών, να αντικαταστήσουμε την αρχή της, ε, του φτηνότερου, του χαμηλότερου κόστους προς εκείνη του πιο βιώσιμου και οικονομικά συμφέροντος κόστους είτε δηλαδή θέτοντας έναν καλύτερο ορισμό των κριτηρίων, να σκεφτούμε δηλαδή εάν είναι, αποδεκτή, εάν είναι αποδεκτός ο τωρινός ορισμός και το σκεπτικό πίσω από αυτόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν κατά πολύ στις τροπολογίες και θα ήθελα να τους ζητήσω να μας πούνε αν είναι αποδεκτές ε, εάν χρειάζονται επεξηγήσεις και την άποψή του σε αυτό. Με άλλα λόγια, με τα χαράς, ε, να θέσουμε ίσως μια, μια ημερομηνία συζήτηση στο Στρασβούργο έτσι ώστε να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Λίγοι μόνο τομείς χρειάζονται συμβιβαστικές τροπολογίες. Οι περισσότερε τροπολογίε χρειάζονται απλά έτσι μια εξετάση, μια ίσως συμπλήρωση, έτσι ώστε να τις ε, παρουσιάσουμε συνολικά και να τις εξετάσουμε και να δούμε δηλαδή αν χρειάζονται κάποιες μικρές προστίκες ή κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ορίσουμε μια ημερομηνία στο Στρασβούργο έτσι ώστε να εξετάσουμε το θέμα λεπτομερώς. Οι περισσότερες τροπολογίες που καταθέσατε μπορούν να γίνουν αποδεκτές από εμένα, διότι είτε ζητούν έναν επακριβές ορισμό, είτε κάνουν μικρές προσθήκες και τροποποίησεις. Όσον αφορά τη γενική στάση στις τροπολογίες, προσπάθησα προσωπικά να διατυπώσω όσο το δυνατόν ακριβέστερους ορισμούς, διότι ε, σε ορισμένους τομείς η εθνική νομοθεσία μπορεί να καλύψει το ζητούμενο. Και ορισμένοι τομείς υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το εξέτασα διεξοδικώς εάν εδώ Ε, εδώ πρέπει να εξετάσουμε τις ε, διαφορές ανάμεσα στο ποινικό δίκαιο και στο εμπορικό δίκαιο στα εκάστοτε κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ένας ε, ευρωπαϊκός ορισμός δεν έχει κάποια προστιθέμενη αξία. Καλύπτονται από τις εθνικές νομοθεσίες. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο μας αφορά στον τομέα των μεταφορών είναι το ερώτημα των ε, υπεργολαβιών. Εδώ εμείς πρέπει, εξετάζοντας τις τροπολογίες, να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι να ληφθούν υπόψη οι μικρές επιχειρήσεις ως υπεργολάβοι και να συμμετέχουν στις ε, δημόσιες συμβάσεις υπό προποθέσει. Εάν η διαχείριση του συνολικού έργου, και τώρα δεν θέλω να αναφερθώ εξε, ε, ακριβώς στο γερμανόφωνο δίκαιο, αλλά για παράδειγμα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επί πολλά χρόνια ανα, πρέπει να πρέπει να περιμένουν τις, να αναλάβουν κάποια υπεργολαβία από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι κανονισμοί πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι κανονισμοί της ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων. Να δούμε τι θα γίνει με τις πληρωμές, αν γίνεται προκαταβολικά πληρωμή ή μετά την ε, παράδοση του έργου. Να βρούμε δηλαδή και εδώ μια ισορροπία διότι πρακτικά είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και είναι ε, ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Και πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν εδώ στις ρυθμίσεις αυτές και τα συμφέροντα των υπεργολαβιών, των υπεργολάβων. σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλές και διαφορετικές πρακτικές στα κράτη-μέλη. Να σας πω για ορισμένες τροπολογίες συγκεκριμένα για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα. Μπορώ να δεχτώ τις περισσότερες τροπολογίες που καταθέσατε, αγαπητοί συνάδελφοι, και ελπίζω κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων να προχωρήσουμε σχετικά ε, γρήγορα. Η Επιτροπή επί της ουσίας θα καθυστερήσει λίγο με την ε, σύνταξη του σχεδίου και εμείς μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ε, σύντομοι λοιπόν. Όμως θα σας κρατήσω ενήμερους για τις νεότερες εξελίξεις στις, στο σύνολο των επιτροπών που ασχολούνται με τη συνάψη δημόσιων συμβάσεων. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω τις τοποθετήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λίχτενμπεργα. Έχω εδώ τους ε, δύο σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Κούν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σήμερα εκπροσωπεύω τον συνάδελφο Κέβιτς και θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω εγκάρδια για αυτήν την εξαιρετική συνεργασία. Ελπίζω στην ε, επόμενη συνεδρία στις Βρυξέλλες και στο ε, Στρασβούργο να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο για να εξετάσουμε τις επιμέρους τροπολογίες και να δούμε εάν ε, μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια γενική γραμμή ή να εξετάσουμε τις ε, επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, σίγουρα το δίκαιο που αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις ε, καθορίζεται πολύ έντονα από τα εκάστοτε κρατημέλη, τα οποία αναλαμβάνουν και την ευθύνη και είναι ευθύνη τους. Και αυτό το θεωρώ λογικό που προτείνατε. Επίσης, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα όσο τον, όσον αφορά στον τομέα της υποδομής, της, των ε, επενδύσεων ε, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Να προσέξουμε στον προϋπολογισμό να ισολογήσουμε κάπως το ζήτημα των ε, δημοσίων συμβάσεων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Να εξετάσουμε τα επιμέρους ζητήματα, να δούμε τον, ε, το χρονοδιάγραμμα των υποδομών, το χρονοδιάρκειας, να δούμε αν χρειάζονται επενδύσεις στον τομέα αυτό. Τα κριτήρια τώρα για την συμμετοχή των ε, αναδόχων στις ε, προκηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις είναι και αυτό κάτι το οποίο χρειάζεται ξεκάθαρο ορισμό και αυτό είναι το δικό μας έργο. Ε, να δούμε τι γίνεται με το dumping, με την ε, πιο συμφέρουσα οικονομικά ε, πρόταση, όπως είπατε κι εσείς, ε, να κοιτάξουμε το κόστος που θα έχει στο μέλλον, τις συνέπειες, να μην κοιτάμε μόνο για την φτηνότερη λύση, Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές όταν προβλέπεται ένα έργο διάρκεια 30 ετών, πολλές φορές με τη φθηνότερη δυνατή λύση, μετά από 10 χρόνια έχουμε πρόβλημα. Όσον αφορά τον όγκο, τον συνολικό όγκο των ε, προκηρύξεων, πρέπει επίσης να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε ποιες επενδύσει Ποιες, ποια μεγάλα έργα πρέπει να... Ε, ποια μεγάλα έργα χρήζουν ε, ε, περιφερειακών συμβάσεων και ποια πρέπει να γίνουν σε κοινοτικό επίπεδο από κοινοτικούς φορείς. Έτσι, έτσι ώστε να επέλθει ησυχία στον τομέα των επενδύσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Περιμένω την κυρία Λαϊέλα. Σας ευχαριστώ πολύ, γι' αυτό παίρνω το λόγο τώρα. Μάλιστα. Όντως, ένα μεγάλο σημείο των δημόσιων συμβάσεων για την ενιαία αγορά στηρίζεται στην εμπειρία, στηρίζεται στο, στο ερώτημα της εναρμόνισης, να δούμε τι θα γίνει με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορούν εκείνες να συμμετέχουν, ώστε να μην υπάρχουν ε, αδικίες και ανισότητες στην ανάθεση. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για, το, για την εξαιρετική δουλειά σας και ε, αναμένω με αγωνία να δω τι μπορούμε να προσθέσουμε, τι μπορούμε να τροποποιήσουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Πραγματικά ρυθμίσατε πολύ, ε, πολλά πράγματα και πιστεύω ότι γενικά ακολουθούμε μια πάρα πολύ καλή γραμμή και γενικά με τον όλο φάκελο είμαι απόλυτα σύμφωση, σύμφωνη και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ ε, για την επικείμενη συνάντηση στο Στρασβούργο ώστε να δούμε τις επιμέρους τροπολογίες και πιστεύω πως είναι ξεκάθαρο ότι όλοι μας, ο καθένας από εμά θα ψηφίσει μαζί με τους συναδέλφους των Επιτροπών επί της ουσίας. Θα ψηφίσει, για παράδειγμα, στην Επιτροπή ΙΝΚΟ, η οποία έχει και την εμπειρία και έχει και ένα ευρύτερο φάσμα και σίγουρα είναι πολύ καλά ενήμερη για τις λογικές αλλαγές, λογικές τροπολογίες. Η δεύτερη ε, γνωμοδότηση για το δίκαιο του τομέα των μεταφορών είναι και αυτό ένα σημαντικό σημείο. Όπως είπε και ο κύριος Κούν, το ζήτημα των υποδομών είναι κάτι που θα έχει μεγάλη διάρκεια στην εξέτασή του. Αναμέναμε αρχικά τέσσερα χρόνια, όμως παρατάθηκε η διάρκεια σε έξι χρόνια. Γνωρίζω ότι ενημερώθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες και ξέρω επίσης ότι ορισμένοι ζήτησαν να έχει όριστη διάρκεια η εξέταση του ζητήματος ε, αυτού. Γνωρίζουμε όλοι ότι το ζήτημα των υποδομών είναι κάτι χρονοβόρο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δίκτυα διευρωπαϊκών μεταφορών. Πολλές φορές μας φαίνεται πως δεν έχει τέλος, όμως καλό είναι να θέσουμε ένα όριο, παράδειγμα αυτά τα έξι χρόνια, να εξετάσουμε, όπως είπε και ο κύριος Κούν, το κόστος, να μην ξεπερνάτε το όριο του 4%. Αν και αυτό μου φαίνεται κάπως υψηλό, η πρόταση για την αύξηση στο 15%. Έπειτα η υποχρέωση κατάθεσης ε, αποδεικτικών στοιχείων. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να δούμε. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα σιδηροδρομικά δίκτυα, ε, έχουν ένα έχουν κάποιο, ε, στο θέμα των σιδηροδρομικών δικτύων υπάρχει, υπάρχουν μειονεκτήματα εάν δεν αναμειχθούν και οι ιδιωτικοί φορεί. Αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτά είχα να πω και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τιπάκελ, πιστεύω, ελπίζω οι φιλελεύθεροι να μην έχουν πρόβλημα που τους αντιπροσωπεύετε εσείς και, να... θα, θα, θα μιλήσει και ο συνάδελφός σας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Κατέθεσα προσωπικά μία τροπολογία, την εξαίρεση. Αυτή που αφορά ορισμένες κρατικές εταιρείες. Και η κατάσταση είναι σοβαρή, είναι δυσεπίλητη, διότι έχουμε πολλές τέτοιες κρατικές εταιρείες οι οποίες σε μια απορριθμισμένη αγορά είναι ενεργές. Επομένως, θα πρέπει αυτές να μην συμμετέχουν στους ε, διαγωνισμούς και για λόγους ανταγωνισμού και για άλλους. Από την άλλη μεριά, αυτές συνεχίζουν και είναι διοκτησία του κράτους. Επομένως, δυνατόν να έχουν και την πίτα ολάκια και το σκύλο χορτάτο. Να λένε ότι είμαστε σε την αγορά, από την άλλη ότι έχουμε τα πλεονεκτήματα της κρατικής διοκτησίας και να συμμετέχουμε έτσι στους διαγωνισμούς. Είναι δύσκολη αυτή η προβληματική να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία πάντως για κάποιους ε, κλάδους. Μπορεί να δείξουν περισσότερη κατανόηση, ας πούμε, στα, για τα, τα, τα υπηρεσίες. Εκεί κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα, όμως για, άλλες, ε, για, άλλους, για, κλάδους δεν ισχύει αυτό. επομένω το να δώσουμε μια γενική εξαίρεση για όλες αυτές τις εταιρείε σε μια προθυμισμένη αγορά, αυτό είναι υπερβολικό, είναι ακραίο. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι δύσκολη η, η, απάντηση που πρέπει να δοθεί. Καλά. Ε, μέσω των μετόχων, εκεί που το κράτος έχει την πλειοψηφία των μετοχών, ίσω να πρέπει να το δούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Να δούμε. Πάντως, είναι μια από πιο σοβαρές συζητήσεις που οφείλουμε να κάνουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, λέει ο κυρία Γιάλα Σέντερ. Λυπούμε κύριε Πρόεδρε. Είχα μια, μια συνεδρίαση, δεν ήρθε και το αυτοκίνητο. Λυπούμε. Εγώ θέλω να, ευχαρι... συγχαρώ την συνάδελφο Μπέργερ για την πρότασή της. Ε, εμείς συμμεριζόμαστε αυτήν την συνέστηση ότι χρειάζεται να πάμε προς μία απλούστευση χωρίς όμως να μειώσουμε την αυστηρότητα και τις απαιτήσεις μας. Ε, βέβαια αυτό το οποίο λέει, αναφέρει η κυρία Λίχτεμπέργεν για επάνωδο στις, ε, στους εθνικούς ε, κανόνες Ε, ε, σχετικά με το θέμα του cross-border, να μπορέσουμε δηλαδή να ξεπεράσουμε αυτούς τους εθνικούς κανόνες και λόγω της κατάστασης να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και να γκρεμίσουμε επίσης και τα εμπόδια με όλες ε, τις προδιαγραφές και απαιτήσεις να μπορέσουμε να έχουμε ρήτρε περιφρούρησης προς τρίτες χώρες οι οποίες έχουν από τη μια μεριά κλειστές τις αγορές τους αλλά από την άλλη συμμετέχουν ανοιχτά στην ευρωπαϊκή αγορά. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδες να διατηρήσουμε όλες τις κοινωνικές πτυχές για να αποφύγουμε και το κοινωνικό ντάμπινγκ και να προστατεύσουμε το κοινωνικό κεκτημένο και τις προδιαγραφές ε, και επίσης ε, πρέπει να προσέξουμε ορισμένοι τομείς όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να δίνουν παράδειγμα τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, δηλαδή οι κανόνες που εμείς θα εγκρίνουμε να μην ε, επιβαρύνουν τον δημόσιο τομέα και να μην επωφεληθούν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν αυτό το κομμάτι δημοσίου τομέα από τα καινούργια μέτρα. Ο κύριος Γκρός. Μάλιστα. Θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτό που είπε ε, ο συνάδελφος Ντεμπάκερ. Αυτό το θέμα πραγματικά είναι σημαντικό και είναι και πολύ ενδιαφέρον. Ήδη ασχοληθήκαμε με αυτό και με την αρχή της ε, αμοιβαιότητα στο παρελθόν. Πιστεύω και αν δεν κάνω λάθος ο Επίτροπος Μπαρνιέ παρουσίασε σε σχετικό φάκελο το θέμα αυτό. Πιστεύω πως πρέπει να αποφασίσουμε και να ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και εδώ για μένα η αρχή της αμοιβαιότητας είναι μια μεταβατική λύση Διαφορετικά πρέπει να δούμε την κατεύθυνση στην οποία που θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εύα Λίχτεμπεργ για το ανοιχτό πνεύμα το οποίο επέδειξε. Και περιμένω στο Στρασβούργο να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας στο Στρασβούργο. Εγώ θέλω να αναφέρω την τροπολογία 52, διότι η κρίση πλήττει κατάφορα την τοπική αυτοδιοίκηση και τα όργανα, τοπικά όργανα. Εγώ αναφέρομαι λοιπόν σε αυτήν την τροπολογία για τα τοπικά προβλήματα. Ε, ξέρετε ποιες προσπάθειες εκλεγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να μειώσουν ε, τις ε, δαπάνες τους Οπότε πρέπει να τους ε, διευκολύνουμε και όχι να τους ε, μπερδέψουμε παραπάνω. Θυμίζω το άρθρο 8 του κώδικα των δημοσίων ε, συμβάσεων της Γαλλίας που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συσπήρωση, μία συνένωση, ούτως ώστε να, γίνονται, να συνάπτονται συλλογικέ δημοσίες συμβάσεις. Έτσι όπως αναφέρεται όμως στο άρθρο 35 στην παράγραφο 3, θέλει να ε, φαίνεται να θέλει να απαγορεύσει σε, αυτά τα, σε αυτές τις εισπυρωμένες ε, ενώσεις ε, αγοράς να παρεμβαίνουν στις, συλλογικές, στις αγορές των δημοσίων συλλογικών συμβάσεων. Γιατί ε, πολλές φορές ε, στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούμε να έχουμε έναν τέτοιο οργανισμό αγορών που να θέλει να αγοράσει συλλογικά πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο υλικό. Θα, πρέπει από το κείμενο να βγει ο όρος «σελ» μόνο, δηλαδή ότι μόνο ο οργανισμός ε, ε, συλλογικών αγορών να μπορεί να αγοράζει, αλλά να μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικές δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστούμε τον, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης για τα θέματα της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις πρώτο πρώτο όσον αφορά τις ποσότητες, όσον αφορά τα κατόφλια και τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται. Σας έχουμε επισημάνει ότι έχουμε διεθνείς δεσμεύσεις ως θεσμικά όργανα για τον GPI. Και αυτό καθορίζει και τα κατόφλια για την εφαρμογή των οδηγιών για τους διαγωνισμούς. Επίσης, όσον αφορά την αμοιβιότητα. Κατά πόσο πρέπει να είναι ανοιχτές οι αγορές μας σε τρίτες χώρες. Σας παραπέμπω στο σχέδιο κανονισμού. Προσπαθούμε την προσβασιμότητα λοιπόν για τις τρίτες χώρες. Από το Μάρτιο 2012 ξεκίνησε αυτή η πρόταση και θέλουμε να καλύψουμε και τους διαγωνισμούς. Οπότε και εμείς στην πρότασή μας δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένε διατάξεις από αυτού προς το παρόν. Κυρία Λίχτεμπερκ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα από τα επιμέρους σημεία. Πρώτα όμως μια παρατήρηση που έχει να κάνει και με αυτό που είπε ο κύριος Πέρκα όσον αφορά τις εξαιρέσεις σε συγκεκριμένους τομείς, τις εξαιρέσεις από τις ρυθμίσεις. Αυτό αφορά τις άλλες ε, επιτροπές, όχι Εγώ θα πρότεινα να μην αλλάξουμε κάτι ριζικά. Για παράδειγμα, τα, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Σε άλλα κρατη μέλη είναι απόλυτα δημόσιες, σε άλλες αρχίζουν ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Ε, η λύση που επιλέξαμε είναι να υπάρχει μία γενική προοριθμισμένη υποχρέωση και όσον αφορά τους επιμέρους ορισμούς να υπάρχει περισσότερη αιμοδιότητα στα κράτη-μέλη. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν οριστεί μέσα από κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. Υπάρχουν τα οποία υπόκεινται σε μια γενικότερη ρύθμιση και όλο αυτό, όλο αυτό το δημιουργεί ένα μπέρδεμα σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος και ποιος όχι. Εμένα θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μάθω εσείς τι γνώμη έχετε για το συνολικό τομέα των ε, ταχυδρομικών ε, υπηρεσιών. Προσωπικά προσπάθησα να βρω μία μέση λύση, διότι οι δομές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ διαφορετικές από κράτος σε κράτος για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και γι' αυτό πρότεινα τη συγκεκριμένη λύση στην τροπολογία. Είμαι όμω ανοιχτή για μια επικοδομητική συζήτηση και μάλιστα είναι αναγκαία μια επικοδομητική συζήτηση διότι από τη μία έχουμε συγκεκριμένους τομείς που όπως για παράδειγμα τι δημόσιε συγκοινωνίε ή τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε που έχουν αναπτύξει τις, τα δικά τους ε, συγκεκριμένα πρότυπα και αυτό για μένα δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο εάν αλλάξουμε τα κριτήρια ή ε, εισαγάγουμε νέα κριτήρια στις προϋποθέσεις για τις προκηρύξεις. Ήταν σημαντικό για μένα να γίνει αυτή η διευκρίνηση και θα με ενδιαφέρε πολύ κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας για τις ε, τροπολογίες να συζητήσουμε και να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Θα ήθελα πολύ να μάθω τις γνώμες των ε, πολιτικών ομάδων. Για μένα είναι βασικό ερώτημα και βασικό ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα του κυρίου Κούν για τις ε, προσφορές ε, dumping, για τα όρια και τα ποσοστά. Στα κράτη-μέλη Υπάρχουν εντελώ διαφορετικές πρακτικές. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που οι προσφορές διαφέρουν η μία από την άλλη κατά 50% και σε άλλα κράτη-μέλη κατά 15%. Υπάρχει λοιπόν μία διαφορά και είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα, διότι είναι αρκετά δύσκολο να υπολογίσουμε και να προσπαθήσουμε να φέρουμε σε μία ισορροπία όλε αυτέ τι διαφορέ. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτέ οι περιπτώσει υπόκεινται στις, ε, στην εθνική νομοθεσία. Οι οποίε εθνικέ νομοθεσίε είναι και πολύ διαφορετικέ από κράτο σε κράτο. Τώρα, όσον αφορά τους ε, υποψήφιου ανάδοχου από τρίτε χώρε. Και εδώ έρχομαι στο θέμα της αμοιβαιότητας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε το αν θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτε χώρε. Καταλαβαίνω το, την αμφιβολία σας και σίγουρα είναι κάτι με, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε γιατί οι περιπτώσεις είναι πολλέ. δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Υπάρχουν πολλά επιμέρους ε, ζητήματα. Ε, θα πρότεινα μία να δούμε τι θα γίνει, διότι οι διαπραγματεύσεις ε, προς το παρόν στο ζήτημα της αμοιβαιότητας ε, δεν έχουν ευδοκιμήσει. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια δίκαιη αντιμετώπιση. Δεν είναι εύκολο να αρχίσουμε να το... από την αρχή τελείως. Ίσως μπορέσουμε να βρούμε μια καλή διατύπωση και να τη χρησιμοποιήσουμε ως εφετηρία όμως, όντως, αυτό το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο. Η συνάδελφος Μάισνερ μίλησε για την μέγιστη διάρκεια των υποδομών. Και εδώ οι πρακτικές στα επιμέρους κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικές. Και είναι αναγκαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλογιστούμε τις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν συμφωνώ με μια γενική και απεριόριστη διάρκεια. Διότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ σαφείς. Αυτή λοιπόν η αόριστη διάρκεια για μένα είναι ένα πολύ προβληματικό ζήτημα. Το βλέπω σε πολλές περιπτώσεις σε πολλές χώρες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, οι προθεσμίες είναι υπερβολικά μεγάλες. Και πραγματικά θα επαναλάβω ξανά ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε. Όπως τώρα, όσον αφορά το κόστος, την ανάληψη του κόστους. Εδώ αυτό το ζήτημα είναι πολύ ενδιαφέρον για τα κράτη-μέλη και όχι μόνο για την Αυστρία. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά ένα έργο σε ένα ε, αεροδρόμιο. Και πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που διατυπώνονται οι προκήρυξεις. Δεν έχουν όλες οι αρμόδιες επιτροπές αναπτύξει αυτή τη ρουτίνα, αυτό, αυτό το τελετουργικό όσον αφορά τις προκήρυξεις. Δεν όμως κάνω λόγο για επανακρατικοποίηση. Μην το νομίζετε αυτό. Απλά αυτό που λέω είναι να δούμε τις διαφορετικές πτυχές. Να δούμε τι γίνεται με το, με το ποινικό δίκαιο, ε, για παράδειγμα, στα διάφορα κρατημέλη και να συνδυάσουμε όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια γενική λύση ομπρέλα που να καλύπτει όλους και να χρησιμοποιήσουμε και την αρχή της επικουρικότητας. Δεν έχει κανένα νόημα να διατυπώσουμε ρυθμίσεις για πέντε κρατημέλη και τα υπόλοιπα να μην μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ή να μην τους καλύπτει. Αυτά για την επανακρατικοποίηση λοιπόν. Νομίζω πως ε, απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ξανά να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας και πραγματικά χαίρομαι γιατί η συζήτηση στο Στρασβούργο προβλέπεται έντονη και επικοδομητική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ψηφοφορία προβλέπεται στην Επιτροπή για τις 18 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο με την, της διάταξης. Τώρα περνάμε με, για τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2013. Κυρία Μάισνερ, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ναι, στο σημείο 8... συζητήθηκε με το ΕΛΚ και πρόκειψε μια πρόταση από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Έχω εδώ αυτό το έτοιμο για χωστή ψηφορία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι θα γίνει. Ξέρουμε ότι είστε υπέρ του πρώτου τμήματος και, και κατά το δεύτερο. Αυτό το λέω διευκρινιστικά. Να ψηφίσουμε με ελληνική ψηφοφορία και όποιος δεν έχει ας το πει. Πρώτα απ' τα ποιοι δεν έχουν. Everybody else has got their αυτοί δεν έχουν που είπατε. Και άρα επομένω ε, δηλώσατε το μετά την ψηφορία. Οπότε για να κάνουμε τώρα τον έλεγχο και την ψηφορία με την ελληνική κάρτα και έτσι να ε, δούμε πώς, πώς δεν θα κάνει ζαβολιά το ΕΛΚ και να ψηφίσουν παραπάνω. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Γιος Γκρός. Έχει επιβάλει πειθαρχία στην ομάδα του, βλέπω, οπότε όλα πήγαν καλά. Ξεκινούμε επομένω. με την ε, τροπολογία 66-17. Ντύρο. Πίνε υπέρ. Πίνε κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε παρακάτω τώρα στο 66-18. Τι είναι υπέρ. Τι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66-22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το 21 με την προφορική τροπολογία. Έχετε κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία. Εάν όχι, θα το, ψηφίσουμε μαζί με αυτήν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το 66, 21. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. Απορρίπτεται. Πάμε όμως στο 6601. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66.00. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-1-6. Καλά φορέσατε μας. Έλα μου λοιπόν σήμερα για να το προφέρω καλά. Ξέρετε υπέρ, κατά, αποχές. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ για το 66-16. Ψηφίζουμε. ένα σύνομα πλήν, ψήφισαν όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 66-02 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Στα 6.03, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στα 6.04, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 66-05, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 66.19, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Νομίζω ότι κρίθηκε, αλλά θα γίνει έλεγχο. 66, 19, ένα είναι ένα πλήν, ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 66, 11, υπέρ. Κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε τώρα. Ένα συν, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 66 καταπίπτει, 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-15 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το 66-15. Ένα σύνολο πλήν, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Στα 608. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 609. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. light fridge παρατήρηση, σχόλιο, υπέρ, κατά, αποχές, Λέξη 66-10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και εδώ έχουμε τις τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τρία καταπίπτει. Δύο μερικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 πίπτια το 7 υπέρ κατά Αποχέα εγκρίνεται 8 σε κατά ψηφοφορία το πρώτο το έχει ζητήσει το ΕΛΚ μέχρι εκεί που λέει για να τονώσει την απασχόληση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα Μέχρι που λέει υπογραμμίζει την διευκόλυνση Connecting Europe, έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Στο 8 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίτευε. Το 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 10. Ψηφίζουμε.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 18-20 απορρίφθηκε, για το 17 τώρα. μέρικα τα αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Με την προφορική τροπολογία είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αν ναι, θα ψηφίσουμε και την τροπολογική τροπολογία. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα 21 καταπίπτει και 22. Ποτέ πάμε τώρα στο 23. Το 22 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 22 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. ...25-11, 26-11, 23 υπέρ κατά αποχές, ίδια πλειοψηφία. Τελική τώρα, ψηφοφορία για το σχέδιο ζώματος, ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. 34-1. Τρεις αποχές. Τα συγχαρητήρια στο τέλος. Συγχαρητήρια κυρία Μάισνερ για την ομοθεσή σα. Μάισνερ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Next we have M, sir. I don't know. Παρακάτω τώρα. Is he here? I have to check. But anyway, Just have a two-minute comfort break to rearrange all the top table and uh, two minutes, colleagues. Δύο λεπτό διάλειμμα για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, του ΕΜΣΑ, τον κύριο Μίλη. Κύριε Μίλη, καλώς ήλθατε στην Επιτροπή Μεταφορών. Ο προκάτοχός σας, ο κύριος Ντερόιτερ, είχε έρθει εδώ. Και νομίζω πως ε, η παρουσία του εδώ ήταν πιο συχνή από ορισμένου Ο κύριος Ντερόιτερ πίστευε στην προσωπική ενασχόληση με τις υποθέσεις αυτής εδώ της Επιτροπής Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να συνεχίσετε το καλό προηγούμενο αυτή τη εξαιρετική συνεργασία με τον ΕΜΣΑ και είμαι σίγουρο ότι τα μέλη μας εδώ ανυπομονούν να ακούσουν αυτά που έχετε να πείτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου τιμή Έρχομαι εδώ να συζητήσουμε για, να κάνουμε τελεία απόψεων. Μόλις ανέλαβα στη Λισαβόνα ως νέος εκδοτικός διευθυντής του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ε, κατόπιν τη, του διορισμού μου στις 8 ε, Ιουνίου του 2012 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε ε, για μας ήσασταν βασικός ε, παράγον ε, συνεργασίας γιατί άμεσα διαμορφώσατε την εντολή μας σε μια διαδρομή χρονική που περάσαμε και επίσης εξασφαλίσατε τους αναγκαίους για μας πόρους. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει πετύχει βάσει της γνώσης και βάσει της ε, συνεργασίας. Ε, εντιενώσει δύναμης λέμε. Και αυτό είναι βασικός ε, πυλώνας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κυρίως, να που μιλούμε για παγκόσμιο ανταγωνισμό, ε, η αρχή αυτή, η βασική που προαναφέραμε, είναι βασική προϋπόθεση για βιωσιμότητα, διμερία και ανάπτυξη. Επίσης, όλη μου τη σταδιοδρομία έχω προσπαθήσει να πετύχω αυτούς τους στόχους και θα συνεχίσω και στο μέλλον και θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην ε, θάλασσα, να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Όπως γνωρίζετε, προσωπούμε εμείς μια πραγματικότητα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη γνώμη μου η σωστή διακυβέρνηση είναι το κλειδί για την ε, επιτυχία ή η αιτία της αποτυχίας κάποιου ρυθμιστικής αρχής. Οπότε γι' αυτό και θα πρέπει να σας αναφέρω ότι έχω εκτενή μακρά εμπειρία στα θέματα management όσον αφορά τη θάλασσα. Η ασφάλεια ε, μας, με έχει απασχολήσει λοιπόν η Βόλη Θάλασσα εδώ και 40 χρόνια και έχω δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλα κράτη-μέλη και σε, στην, στην ΕΜΣΑ και στην, στην ε, Οργανισμό Ασφαλής Θάλασσας και νομίζω ότι το έργο που έχουμε επιτελέσει στην ΕΜΣΑ είναι από το 2002 πάρα πολύ αξιόλογο ε, υπό την διοίκηση του κ. Ντερόιτερ και του ικανού προσωπικού. Ήταν αξιοπρόσφυτα τα αποτελέσματά μας και επηρεάσαμε πάρα πολύ ε, στα θέματα τη ασφάλεια και στην Ένωση αλλά και παγκοσμίω. Οπότε και τελικά απολαύουμε σεβασμό σε όλα τα επίπεδα και από όλου του εμπλεκόμενου. Θα θέλω να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και θέλω να πάμε ακόμα καλύτερα όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, την ε, απόσταση στο περιβάλλον και έτσι να έχουμε μια προσταμινή αξία ε, για την Επιτροπή, τα κρατημέλη, τους εμπλεκόμενους και βέβαια και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιο είναι το όραμά μας. Να γίνει η ΕΜΣΑ όλο ένα και πιο γνωστή και στην Ένωση και παγκοσμίω. Το προσωπικό και οι επιδόσεις μας πρόκειται να ωφελήσουν πάρα πολύ την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και τους άλλους εμπλεκομένους. Η εφαρμογή, η θέση σε ισχύ του καταστατικού της υπηρεσίας μας ε, αποδίδει στην Επιτροπή σας πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό θα είναι η βασική πρόκληση Οπότε και εμείς σας διαβεβαιώ ότι πρόκειται να συνεργαστούμε και να βρούμε λύσεις καινοτόμες, δημιουργικές για ό,τι έχουμε να κάνουμε σήμερα και ό,τι θα πρέπει να κάνουμε και αύριο να επιτελέσουμε το έργο μας και επίση πρόκειται να συνεργαστούμε και με τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και με όλους τους εμπλεκομένους για να βρούμε λύσεις βιώσιμες, διαρκείς και τις καλύτερες απλώς πρακτικής. Επίσης, όσον αφορά τη συμβουλευτικό μας έργο, πρόκειται να επηρεάσουμε επί πολύ αποφάσεις, κανονισμούς και νόμους. Επίσης έχουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή πολιτική για θάλασσα, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και αυτό βέβαια θα ωφελήσει και ε, τις εφοπλιστικές εταιρείε. Επίσης, ε, να σας πω πώς βλέπω το προσωπικά την εξέλιξη. Θεωρώ ότι οι καλέ μεταφορέ είναι παγκόσμια σημαντικέ, αλλά και κυρίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολλέ ε, χώρε μέλη εξαρτώνται από, πάρα πολύ από τι καλέ ε, μεταφορέ. Η ασφάλεια στη θάλασσα ε, είναι αντικείμενο ρυθμιζόμενο των IMO, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τι αρμοδιότητέ τη από αυτού και βέβαια συνεργάζεται στην με τον IMO. Οπότε θα πρέπει η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα να ληφθούν υπόψη όσο γίνεται περισσότερο για να μην ξεχνούμε και στη, τα οικονομικά θέματα για τον κλάδο των μεταφορών γιατί έχουμε μια μακρά παράδοση των σκαφών που φέρουν σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε θα πρέπει ο κλάδος αυτός να γίνει βιώσιμος οικονομικά και ανταγωνιστικός στην Ένωση η ΕΜΣΑ θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμη, να έρχεται σε επαφή με επιτροπή, κρατημέλη, του εμπλεκομένου, ούτω ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να εξυπηρετήσουμε τον κλάδο των εργασίων μεταφορών στην Ένωση και έχει αναγνωστεί αξία του οργανισμού μας από όλους τους Αυτό όμως θα πρέπει και εμείς να το ε, αποδείξουμε ότι ισχύει με σκληρή δουλειά, με εξέβρεση λύσεων να είμαστε δυναμικοί, ε, θα πρέπει να προτείνουμε κάποιες λύσεις που θα κάνουν ακόμα πιο φιλοπεριβαλλοντικό τον, τον, τον, τον τομέα της θάλασσας και πιο επικερδή. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι τις οικονομίες των κρατών μελών να ξεπεράσουν την ε, κρίση, να βοηθήσουμε τη βιομηχανία γιατί σήμερα ο τομέας ε, τα φορών απασχολεί 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους και έχουμε ένα σωρό νέους και φοιτητέ ε, που έρχονται για να πιάσουν δουλειά στον κλάδο αυτό και έτσι τους εξασφαλίζεται ένα ρόδινο μέλλον. Ε, δεν μπορούμε να τον βέβαια να ενεργήσουμε από μόνοι μας, απομονωμένοι. Χρειάζεται συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις νομοθετικές αρχές, το Κοινοβούλιο, τις εθνικές αρχές, του άλλου εμπλεκομένους και στον οργανισμό μας με την εμπειρογνωμοσύνη μας θα αναζητήσουμε λύσεις για όλα τα θέματα που θα ανακύψουν. Το κοινοβούλιο γενικά και πιο συγκεκριμένα η επιτροπή σας έχετε πιστέψει μα και έχετε παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αναθεώρηση της εντολής μας. Και θα σας ε, διαβεβαιώσω ότι η ψήφος εμπιστοσύνη μας πρόκειται να αποδώσει καρπούς. Τέλος, οι εσωτερικές δομές και οι διαδικασίες μας θα πρέπει να βελτιωθούν όσο γίνεται και να απαλλαγούμε από τη γραφειοκρατία και θα πρέπει επομένω να δίνουμε την εικόνα μιας ισχυρής ομάδας που έχει δυνατότητες μεγάλες, οπότε και έτσι θα προβληθούμε, θα είμαστε πιο προβλημένοι σε Ευρωπαϊκή και η υπηρεσία μα θα πρέπει να έχει διάλογο υψηλού επίπεδου και αποτελεσματικό με τα κρατημέλη, τα θεσμικά όργανα και του άλλου συμπλεγωμένους. Επίση θα μπορέσουμε να καλύψουμε τι τεχνικέ προκλήσει ε, όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, την πληροφορική, να τα καλύψουμε το πρόγραμμα εργασία μα Δεν θα πρέπει να έχουμε επικάλυψη στο έργο μα με, με άλλα κρατή, με κρατημέλη, τόσο με άλλε υπηρεσίε. και πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε το έργο των κρατών μελών και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να πλαισιώσουμε το έργο των εθνικών αρχών. Θα πρέπει επίσης να είμαστε αισιόδοξοι, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αποτελεσματικοί και θα πρέπει να είναι βιώσιμες και με διαφάνεια οι αποφάσεις μας οι πόροι μας, και οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικότητα για κάθε μας δραστηριότητα. Και τα αποτελέσματα να είναι ορατά και να δίνουν την προσθέμενη αξία σε όλους. Ως συμπέρασμα, σας παραβάνω τα πιο βασικά σημεία που είναι τα εξή. Η αποστολή μας είναι να εξασφαλίζουμε και να βελτιώσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε όλο ένα και περισσότερο σεβασμό ε, όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος του θαλασσίου και θα πρέπει ομένω να είμαστε γνωστοί, προβλημένοι ευρωπαϊκά, παν, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, να έχουμε αποτελεσματική, σωστή χρήση των, ε, των, των πόρων, των δημοσίων, την εμπειρογνωμοσύνη και προσθέμενη αξία και αυτά όλα είναι το πιο σημαντικές έννοιες που πρέπει να έχουμε μπροστά μας. Επομένως θέλουμε καλή εταιρική διακυβέρνηση, να λειτουργήσουμε εύρυθμα και νομίζω ότι αυτά που σας είπα, ε, που σας έδωσαν να καταλάβουν ποια είναι η υποστολή μας και τι θέλουμε να κάνουμε στην έμψα και περιμένω ευχαριστώ τις ε, ερωτήσεις σας και βεβαίως ε, ισχύει πάντα η πρόσκλησή μας για να έρθετε στη Λισαβόνα να μας επισκεφτείτε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιλή. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Μπορούμε να επισκεφθούμε τις ε, υπηρεσίες όπως την ΕΜΣΑ και ελπίζω να το πράξουμε αυτό στο προσεχές μέλλον. Έχουμε μεγάλο κατάλογο ομιλητών. Να αρχίσουμε με τους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Τέσσερα λεπτά ο καθένας και τότε θα έχουμε αρκετό χρόνο για απαντήσεις. Έχουμε κύριε Γκρός, Φλέκενστάιν, κυρία Μάισνερ, κύριος Κράμερ, κύριος Ζήλου για τις ομάδες. Μετά, κύριος Ντεκράντες, αρχικά, θα σας αλλάξω λοιπόν. Κύριε Αλκαντράουι, κύριος Κομουτζάκος, κύριε Σαβάος. Και μετά η κυρία Αϊέλα Σέντερ. Μάλιστα. Κύριε Ντεγκράντες, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κύριε Μίλη, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχόμαστε καλή και επιτυχή εργασία στις νέες αρμοδιότητες που αναλάβατε στις 6 Ιουνίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα υποστηρίχθηκε πάντοτε από το Κοινοβούλιο και υπήρξε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, στενή σχέση μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών και των υπευθύνων του οργανισμού και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και η, η Επιτροπή μας πάντοτε υποστήριξε τις νέες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν σιγά σιγά στον οργανισμό σας. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Αλλά κάτι μετρώει, κάτι σκέφτομαι. Συνέχεια. Ένας από τους λόγους της επιτυχίας της ΕΠΣΑ εδώ στην Επιτροπή μας είναι ότι ποτέ δεν απαγοήτευσε τους ευρωβουλευτές. Ο προκάτοχός σας ερχόταν πάρα πολύ συχνά εδώ στην Επιτροπή μας. Και αυτό αξίζει να το πούμε, διότι υπάρχουν οργανισμοί που πιστεύουν ότι είναι αυτοφύης, ότι μπορούν να ζουν μόνοι τους. και θεωρεί ότι είναι υπόλογοι μόνο στην Κομισιόν. Δεν θα πρέπει οι οργανισμοί να ζουν στο περιθώριο θεωρώντας ότι είναι ε, ε, οντότητες από αυτές. Αυτό αποτελεί λοιπόν, ε, αυτή η διαφορά αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας της ΕΨΑ. Γι' αυτό λοιπόν και η Επιτροπή μας κάθε φορά που ζητήσατε νέες αρμοδιότητες πάντοτε είπαμε ναι. Πρόκειται όμως για μία επιτυχία τεκμηριωμένη σε αυτήν την πρακτική. Ο κύριος Μίλη είπε ότι είναι πολύ σημαντική η αναφορά της Όμη. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Και εμείς σίγουρα θα πρέπει να λειτουργούμε στο πλαίσιο αυτό. Αλλά αν εμείς περιμέναμε όμως μόνο την νόμη να, ε, λαμβάνει, ε, να, λαμβάνει τις, ε, να, λαμβάνει, να δράσεις ας πούμε για τα πλοία με, τις, με, το, το διπλό τείχομα ακόμη θα περιμέναμε. Η ΕΜΣΑ είναι αυτή που αναλαμβάνει τελικά την ε, πρωτοβουλία και αυτό είναι και το κλειδί. Πάντοτε να μπορούμε να, ενεργούμε κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών και να ε, υλοποιούμε τις αποφάσεις της Κομισιόν. Εδώ και κατά την έκθεση του κυρίου Φλενκεστάιν είχαμε μια τεράστια συζήτηση για το ρόλο της ΕΜΣΑ και όπως είπατε αποτελεί μία αναφορά η οποία είναι βασική για τη λειτουργία της. Λοιπόν, τώρα σήμερα είναι η πρώτη σας μέρα. Θέλω να σας επαναλάβω εξ ονόματος της ομάδας μου καλωσόρισες. και να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου και τη σιγουριά μου ότι θα συνεχίσει η ΕΜΣΑ να πληρεί τον όρο της για την, το, το ρόλο της για την ασφάλεια στη θάλασσα και ότι θα έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλέκενστάιν, μην ξεπεράσετε τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζομαι καν τέσσερα λεπτά. Σας καλωσορίζω κι εγώ εκ μέρους της ε, ομάδας μας. Αναφέρθηκε ήδη πάρα πολλές φορές ότι αυτή η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό σας με χαρά και ελπίζουμε να μπορούμε να υπολογίζουμε σε σας και στο μέλλον. Ε, όπως ε, είπε και ο προλαλή σας, ε, είχαμε πολλές επικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ σας, αλλά και με το Συμβούλιο. Ορισμένες από αυτές πήγαν καλά, ορισμένες δυστυχώς όχι και τόσο καλά, διότι δεν μπορούσαν όλα τα κράτη-μέλη να πείσουν τους αντιπροσώπους τους για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Διατυπώθηκαν διαφορετικές ε, θέσεις για το πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ε, θέσεις της, ε, του ΕΜΣΑ. Είδαμε ότι όταν αλλάζει η νομική υπόσταση, για διάφορους λόγους σε κάποιο κράτος μέλος, τότε υπάρχουν... υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση. Εμείς ακόμα και αν βρισκόταν έτσι σε θελοντικό επίπεδο, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανταλλαγή καλών πρακτικών, μια ανταλλαγή κατάρτισης και εμπειριών. Και όσον αφορά την ασφάλεια των ε, σκαφών μας, Ελπίζουμε να μπορέσουμε να θέσουμε σαφείς προθιαγραφές και σε αυτό ελπίζουμε να συνεισφέρει σημαντικά και ο ΕΜΣΑ. Και για μένα αυτό δεν ε, αφορά μόνο τα σκάφη που δραστηριοποιούνται στο κέρας της Αφρικής, αλλά και σε, άλλους, ε, και σε άλλες περιοχές. Ε, κάτι τελευταίο Ε, κύριε Μπάουερ δεν είναι εδώ και θα ήθελα να σας το πει η ίδια. Αλλά ελπίζουμε να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στον ΕΜΣΑ. Κάτι που θα ήθελα να πω κλείνοντας. Αρμοδιότητες χρειάζονται Περισσότερες αρμοδιότητες χρειάζονται, δυστυχώς όμως δεν έχουμε και περισσότερες δυνατότητες για αύξηση του προϋπολογισμού. Έχουμε πολύ περιορισμένα μέσα. Μόλις ψηφίσουμε στο τέλος της χρονιάς, ελπίζω να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα που επιθυμούμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας υποστηρίξουμε και με τα μέσα που χρειάζονται και θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε αυτά τα μέσα που θα θέσουμε στη διάθεσή σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τους φιλελεύθερους η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Μίλη, εδώ είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και που μας παρουσιάσατε. Για μας ο ΕΜΣΑ είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Φλέκενστάιν που μίλησε για το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών. Όντω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι γενικότερα ο ναυτιλιακός τομέας πάσχει σε αυτό το θέμα και σε γενικές γραμμές όμως ε, είναι σημαντικό ο ΕΜΣΑ να ηγηθεί στον τομέα της ασφάλεια. Λίγο πριν έρθετε μιλήσαμε για τον, ε, ψηφίσαμε τον προπολογισμό του επόμενου έτους και μάλιστα και για τον ΕΜΣΑ γιατί περιμένουμε πολύ περισσότερα πράγματα από τον ΕΜΣΑ. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας και σας δώσαμε περισσότερα χρήματα για την ε, κατάρτιση προσωπικού. Τουλάχιστον αυτή εδώ η Επιτροπή προσπάθησε και είναι στο πλευρό σας. Εγώ προσωπικά είμαι, ε, γνωμο, ε, είμαι υπεύθυνη για την ε, θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι συγγήτρια και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ένα τομέα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τι επόμενε γενιέ. Και είναι επίση πολύ σημαντικό να προσέξουμε και το ζήτημα, το περιβαλλοντικό ζήτημα και την προστασία του περιβάλλοντο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έγινε μια αβαρία στον Βόρειο Ατλαντικό. Ίσως δεν το πρόσεξαν πολύ. Ένα γερμανικό πλοίο που ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη προς τον Bremerhaven στη Γερμανία. Ε, έγινε μια έκρηξη και πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Φλέκενστάιν, είχαμε ε, ζητήσαμε βοήθεια, όμως δεν λειτουργήσε το σύστημα. Γενικώ αυτό το σύστημα έχει προβλήματα σε διεθνές επίπεδο στο, στην ε, βοήθεια των γειτονικών χωρών. Υπήρχαν δυνατότητες να έχουμε βοήθεια από τα γειτονικά κράτη, όμως στην πράξη αυτό που έγινε είναι ότι η Γερμανία ανέλαβε μόνη της αυτό το έργο και πραγματικά είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τομέα της συνεργασίας για την ασφάλεια των σκαφών. Η οδηγία της Επιτροπής 17 από το, από το 2007 αναφέρεται σε αυτό. Ακόμα έχουμε ζητήσει μία εξέταση, δεν έχουμε όμως ακόμα τα αποτελέσματα της μελέτης του τι γίνεται σε περιπτώσεις αφαρίας γιατί πραγματικά δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα βελτιωθεί αυτός ο τομέας στο μέλλον, πώς θα περιοριστούν οι κίνδυνοι. Πρέπει να εντοπίσουμε βέβαια τους κινδύνους αυτούς και, για να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε και ελπίζουμε μαζί με τον ΕΜΣΑ να εργαστούμε προς αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Μάισνερ, ο κύριος Κράμερ για τους πράσινους τώρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ με τη σειρά μου και πραγματικά μου κάνει μεγάλη έκπληξη η, ε, η αναφορά στο γερμανικό πλοίο. Έγινε στις 6 Ιουλίου το πλοίο Φλαμίνια τυλίχθηκε στις φλόγες και στις εργασίες πυρόσβεσης έχασε τη ζωή του ένας ε, ναύτης στα μέσα Ιουλίου. Τότε έγινε το ατύχημα, ατύχημα καμία χώρα δεν ήταν στη θέση να παράσχει βοήθεια, σωστική βοήθεια όταν έγινε αυτό. Και κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Μέχρι τώρα αυτό είναι άγνωστο. Έπρεπε το πλοίο να οδηγηθεί στο γερμανικό λιμάνι, ενώ θα μπορούσε να πάει κάπου πολύ κοντύτερα, αλλά έλειπε, έπασχε αυτό το θέμα. Σε αυτό οι διεθνείς οργανισμοί απέτυχαν και να σας ρωτήσω, ήσασταν εσείς αναμειγμένοι σε αυτό. Κάνατε κάτι γι' αυτό. Οδηγήσατε το πλοίο στο πλησιαστερό λιμάνι, ζητήσατε βοήθεια. Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Αλλά επειδή το πλοίο δεν είχε, σημαία είχε γερμανική σημαία και δεν ήταν σημαία άλλων κάποιου κοντινού κράτους, δεν, δεν, δεν υπήρξε καμία βοήθεια και είχαμε, χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Πώς αντιδράσατε, πώς αντέδρασε ο ΕΜΣΑ και ποιες ήταν οι δικαιολογίες εκείνων που αρνήθηκαν να παράσχουν βοήθεια. Τι χρειάζεστε εσείς, ποιο ρόλο θέλετε, ποια είναι τα εμπόδια που έχετε για να, πραγματοποιήσετε το έργο σας. Είστε πραγματικά ένας διεθνής οργανισμός ή υπάρχει κατακαιρματισμός σε μικρά εθνικά συμφέροντα. Πρέπει πραγματικά να δούμε την πραγματικότητα με γυμνό φαλμό, η οποία δουμε την πραγματικοτητα με γυμνο η οποια ειναι και σκληρή πολλές φορές. Πραγματικά, δείτε τι έγινε. Και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να έχω κάποια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας πείτε σε τι στερήσατε. Δεν ήταν εθνική ευθύνη της διάσωσης του πλοίου. Ήταν ευρωπαϊκή ευθύνη. Και αυτό που έγινε είναι ότι έμεινε, αποδόθηκε η ευθύνη σε ένα κράτος, το κράτος που είχε, τη σημαία του οποίου είχε το πλοίο. Έγινε αυτό πριν από έξι εβδομάδες. Και τι έγινε, το είπαν ότι το πλοίο πρέπει να πάει στην ε, ακτή και έπρεπε μάλιστα να περάσει από το, κομμάτι, το γερμανικό κομμάτι της ε, Βόρειας Θάλασσας. Αλλά πραγματικά ήταν μεγάλη καταστροφή. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή ναυτιλία και καταστροφή στα, των τελευταίων χρόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς δεν έμαθε τίποτα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ Μάικλ. Κύριε Γκρός, τρία λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καλωσορίζω τον Διευθυντή για το, για το διορισμό του και εύχομαι να συνεργαστούμε καλά. Ο ο οργανισμός σας είναι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ καλά και ελπίζω ότι κατά τη θητεία σας και θα συνεχίσει να λειτουργεί εξίσου καλά. Εγώ ήδη έθεσα διάφορα σημεία και θα ήθελα να προσθέσω ακόμη ένα σχετικά με το θέμα των σταδιοδρομιών και της εργασίας ε, στη θάλασσα για τους νέους. Φυσικά για να ενθαρρύνουμε τους νέους να γίνουν ναυτικοί χρειάζεται να δώσουμε εκπαίδευση και κίνητρα για αυτή την εκπαίδευση. Εσείς ε, στον οργανισμό σας για την ασφάλεια στη θάλασσα θα παρέμβετε με πρωτοβουλίες ε, για να προσελκύσετε τους νέους προς αυτόν τον τομέα Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, θα σας ευγνωμονούσα. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία με τη σειρά μου στο έργο που αναλαμβάνετε. Υπόθηκε ήδη και το επαναλαμβάνω και εγώ ότι η Επιτροπή αυτή έχει δώσει την υποστήριξή της προς την ΕΜΣΑ. Μια υποστήριξη σταθερή στο βάθος του χρόνου και έχουμε δώσει την υποστήριξή μας επειδή πιστεύουμε ότι η δράση της ΕΜΣΑ μπορεί να έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια που κάνει η Ένωση να διατηρήσει και να ενισχύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει παγκοσμίω η ευρωπαϊκή ναυτιλία. Μια ναυτιλία ασφαλής, ποιοτική και ανταγωνιστική. Ε, θα ήθελα να σας πω βεβαίως ότι αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις ότι η υποστήριξη αυτή δεν είναι μια λευκή επιταγή. Ο βαθμός υποστήριξης που δίνουμε στην ΕΜΣΑ είναι βεβαίως, όπως σε όλους τους οργανισμούς, μην παρεξηγηθώ γι' αυτό, ε, δεν είναι μια λευκή επιταγή. Ο βαθμός υποστήριξης που δίνουμε είναι ε, ανάλογος και συνδεδεμένος με τον βαθμό της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Ε, μέχρι τώρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Με αυτή την ευκαιρία που σήμερα είσαστε εδώ για να μας ενημερώσετε, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα για να έχω την αντίδρασή σας. Ε, όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο θα απασχολήσει ε, το Κοινοβούλιο και γενικότερα την Ένωση ε, η, οδηγία για την τροπο, η συζήτηση για την τροποποίηση της οδηγίας του 2009 ε, σχετικά με την έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας. Ε, εκεί υπήρξε μια συζήτηση που έγινε στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και εκφράστηκε μια ενδιαφέρουσα ιδέα και θα ήθελα να έχω την αντίδρασή σας αυτήν. Ε, η ιδέα είναι ότι επειδή ο, ο έλεγχος που θα γίνεται από το κράτος λιμένα θα γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, δεν, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αρκετοί επιθεωρητές που έχουν αυτή την τεχνική γνώση, την πλήρη τεχνική κατάρτιση, για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη συζήτηση που έκανε ε, κατέγραψε μια ιδέα ώστε η ΕΜΣΑ να βοηθήσει ή εν πάση περιπτώσει να αναλάβει την, να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατάρτιση των επιθεωρητών πριν την έναρξη ε, της ισχύω της Σύμβασης για την Αυτική Εργασία, ώστε να είναι εγκαίρος σε θέση οι επιθεωρητές να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους από αυτή τη Σύμβαση ελέγχους. Ε, και ε, καλείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η ΕΜΣΑ, και τα κράτη που έχουν προσυπογράψει το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων, το MOU, ε, για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, να προωθήσουν δυναμικά το ζήτημα της κατάρτισης των επιθεωρητών για το σκοπό αυτό. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς σε πρώτη ανάγνωση αντιμετωπίζετε αυτή την ιδέα και εάν ε, στον τρέχοντα προϋπολογισμό και με τις οικονομικές δυνατότητες που ήδη υπάρχουν στην ΕΜΣΑ θα μπορούσε ενδεχομένως να καλυφθεί μια τέτοια αποστολή από την πλευρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σαβράμα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, συγχαρητήρια, αλλά και πολύ καλή τύχη στο τόσο δύσκολο έργο σας, κύριε. Θα ήθελα τώρα να πούμε δύο λόγια για την περιοχή της Βορειοελτικής θαλάσσης. Έχουμε βέβαια στρατηγικό ρόλο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ε, θάλασσα Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε όχι μόνο για την περιοχή αλλά πιο συγκεκριμένα για τον κόλπο της Φινλανδίας. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι εδώ στην Επιτροπή δεν είχαν την ευκαιρία να προσέξουν τι γίνεται σε αυτή την τόσο μικρή λιμνούλα ούτως υπήν, γιατί είναι πάρα πολύ ε, στενός αυτός ο κόλπος και έχει πάρα πολύ κυκλοφορία εκεί που ε, αυξάνεται εκθετικά. Επίσης η Αγία Πετρούπολη ε, χρησιμεύει για, σαν εξαγωγικό λιμάνι της Ρωσίας, οπότε η κίνηση εκεί, η κυκλοφορία εκεί, η ναυσιπλοεία εκεί γίνεται απίστευτη σε ποσότητα. Οπότε για πέστε μας τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κοινοβούλιο κατά τη γνώμη σας. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την να την ασφάλεια της Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Μίλη. Σας συγχαίρω κύριε Μίλη για το διορισμό σας. Ελπίζω να πετύχετε στο έργο σας. Εγώ θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Δεγκράντες Χρειάζεται η συνεχής παρουσία της ΕΜΣΑ για να συνεχιστεί δηλαδή και η παράδοση εδώ στο Κοινοβούλιο και ο αποτελεσματικός ε, διάλογος και συνεργασία. Εσείς ε, έρχεστε με... Ε, αναλαμβάνετε αυτό το έργο με τεράστια εμπειρία, εμπειρία συσσωρευμένη από τη δουλειά σας στα λιμάνια ε, έρχεστε από το χώρο της Βαλτικής. Ποια είναι όμως η εμπειρία σας με την Μεσόγειο. Το θέμα της οδηγίας ε, ε, για μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Εμείς η Μεσόγειο δεχτήκαμε το, το είδαμε με κακό μάτι το θέμα των ε, λιμανιών γιατί είχαμε την αίσθηση ότι ετέθη ένας ανταγωνισμός μεταξύ των λιμανιών του Βορρά και των ε, λιμανιών του Νότου. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει και ένα fair play μεταξύ της εμπειρίας σας ε, στον χώρο της Βόρειας Θάλασσας ε, και αυτό το fair play θα πρέπει να είναι εξίσου καλό και για τα λιμάνια της Μεσογείου που έχουν τεράστια δυναμική και είναι ανοιχτά ε, στις ε, χώρες της Βόρειας Αφρικής με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης, για τους ναυτικούς, εσείς τι σκέφτεστε σχετικά με τις συνθήκες ζωής τους Έχουμε όλο ένα και λιγότερους Ευρωπαίους ναυτικούς. Κρατάμε μόνο τους ε, Ευρωπαίους, ε, ε, μάλλον συγγνώμη, περιορίζονται και οι Ευρωπαίοι πλοίαρχοι στα πλοία μας γιατί οι συνθήκες γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες. Μήπως θα έπρεπε η ΕΜΣΑ να προωθήσει έναν συντονισμό, συντονισμό για την βελτίωση της ζωής αυτών των ναυτικών, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες και να ξεκινήσει και εκστρατείες πληροφόρηση σε τέτοια φάση, δηλαδή κρίσης απασχόλησης κλπ. Οι νέοι Ευρωπαίοι να δούνε πόσο θελκτική μπορεί να είναι η ζωή στο ναυτικό. Για το θέμα της πειρατείας και της ε, τρομοκρατίας, τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει ο οργανισμός είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για το οποίο πρέπει να αναπτύξει ιδιαίτερα τις δυνάμεις της Ευρώπη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, αναφέρθηκε πάλι το ζήτημα του εμπορίου και να τονίσω την ανάγκη να φέρουμε τους Ευρωπαίους πολίτες στον ναυτιλιακό τομέα. Ως αξιωματικούς σε εμπορικά πλοία μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν ανεβαίνει στη γέφυρα ενός πλοίου και βλέπεις Ευρωπαίους αξιωματικούς, με το που κατέβησε όμω από τη γέφυρα, του ψάχνει με το κιάλι. Όντω υπάρχει λοιπόν μία ανάγκη γι' αυτό. Έπειτα, το επόμενο ζήτημα έχει σχέση με αυτό που ανέφερε ο κύριος Κράμερ, με το ατύχημα του γερμανικού πλοίου, το δυστύχημα μάλλον. Είναι δύσκολο. Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε πρώτον το ρόλο σας και δεύτερον να κάνουμε τα κρατημέλη να τον αποδεχτούν. Όπως και οι συνάδελφοί μου και εγώ το βρίσκω αποτρόπαιο ότι ένα πλοίο που είχε πρόβλημα αφέθηκε στην τύχη του και δεν το βοήθησε κανείς να φτάσει σε ασφαλές λιμένα. Κανένα άλλο κράτος δεν ενδιαφέρθηκε και αυτό είναι, είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο όλων των κανόνων ναυτιλιακής δεοντολογίας, όλων, όλων των παραδόσεων που είχαμε στη θάλασσα όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει όντω μεγάλο θέμα με αυτό το γερμανικό πλοίο και πραγματικά θα με ενδιαφέρει η απάντησή σα. Δεν υπάρχει κάποιο ε, από την Επιτροπή αρμόδιο εδώ, αλλά πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω όπω ένα Φίλιπ να το μεταφέρει στην Επιτροπή και να του ζητήσει να απαντήσουν και να πούν. Να τοποθετηθούν γι' αυτό. Επίση, κάτι άλλο που με απασχολεί είναι το γεγονός ότι... Θα σας δώσω ένα παράδειγμα του προβλήματος που ξέρετε πώς αντιμετωπίζουμε. Ήμουν, είχα παρευρεθεί σε ένα συνέδριο των ε, σχετικό με την ναυτιλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο αντιπρόσωπο μιλούσε για την ασφάλεια στην θάλασσα και για όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε στο ναυτιλιακό τομέα για να επιτευχθεί αυτό. Και κατά τη μισή ώρα που μιλούσε ποτέ δεν ανέφερε ούτε μία φορά την, ε, τον ΕΜΣΑ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε μία φορά. Αμέσως μετά πήρα το λόγο και τους έθιξα το θέμα αυτό. Και όλοι χειροκρότησαν τότε και είπαν πραγματικά γιατί δεν, αναφέρθηκαν η ΕΜΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει καρφωθεί αυτό στο κεφάλι τους και πραγματικά με ανησυχεί. Γιατί δεν είναι μόνο βρετανικό το ζήτημα, υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η αδιαφορία και πραγματικά εάν αλλάξει η νοοτροπία τότε θα θα βρεθεί λύση. Τότε θα έχει αποφευχθεί και το πρόβλημα, το δυστύχημα αυτό με το γερμανικό πλοίο. Είναι όντω ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό που σας ζητώ να αναλογιστείτε είναι πραγματικά να πιάσετε μία-μία τις ναυτιλιακές αρχές στα κρατημέλη με, αναλόγως με το που υπάγεται η καθεμία, δεν υπάγονται όλες στον ε, ίδιο φορέα, αλλά να τους πιάσετε, να τους συγκεντρώσετε όλους και να τους πείτε ότι εδώ αυτό είναι το έργο σας. Αυτό πρέπει να κάνετε, είστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το κάνετε. Κιθ, θέλεις να πεις κάτι, δεν ήξερα ότι ζήτησε το λόγο, αλλά έχεις τώρα το λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Μπράιεν. Νόμισα πως δεν με είδες. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη νέα σας δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθούμε στη Λισαβόνα. Είχα την τύχη να πάω πέρυσι και να δω τα νέα κεντρικά σας γραφεία και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο επαγγελματισμός σας και η εμπειρία των συνεργατών που ήταν προφανής. Προσωπικά και μιλώντας εκ μέρους των συναδέλφων μου, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός ε, ε, στην, ε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας, αλλά για μένα το θαλάσσιο περιβάλλον δεν αναφέρθηκε αρκετά. Αναφέρθηκε αλλά όχι αρκετά. Πολλά είναι τα ερωτήματά μου. Το κύριο όμως ερώτημα είναι εάν μπορείτε να μας δώσετε μία περιγραφή του πώς η ΕΜΣΑ θα προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην θάλασσα. Και θα ήθελα να μου απαντήσετε εάν θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή στήριξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, ναι, έχουμε κάποιον από την Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω από τον κύριο Μπόσουμ να μα πει, μη ξέρετε το όνομα του γερμανικού πλοίου Φλαμίνια. Το πλοίο Φλαμίνια λοιπόν. Γιατί πραγματικά, για να είμαι ειλικρινή, κύριε Μπόσουμ, αυτό είναι κάτι που οφείλετε να μα απαντήσετε. Έχετε να μα δώσετε κάποιε εξηγήσει. Κύριε Μάλιστα, με τα χαράς. Καλημέρα. Δεν έχω προετοιμαστεί να σας εκθέσω με λεπτομέρειες το περιστατικό του πλοίου Φλαμίνια, αλλά θα μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία. Φυσικά ήταν τραγικό δυστύχημα και πραγματικά αυτό θέτει το θέμα της ασφάλειας των ε, κοντέινερ στην θάλασσα και πραγματικά αυτό το ερώτημα πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργά ε, συντόνισε τη δράση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ερωτήματα των κυρίων Κράμερ και της κυρίας Μάισνερ για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτι που απασχόλησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως το ερώτημα της αρμοδιότητας της ΕΜΣΑ. Και λοιπόν ε, θεωρήθηκε επίγον να ληφθεί μια απόφαση. Οδηγεί 2005 κάθετος 9 ρυθμίζει το ζήτημα, όπως είπε και η κυρία Μάισνερ, αλλά να πω ότι αυτή η οδηγία δεν δίνει ξεκάθαρα, δεν προβλέπει ε, αποκλειστικέ αρμοδιότητε ούτε για την ΕΜΣΑ ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να επεξεργάζεται την οδηγία. Διατυπώθηκαν κάποιες προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν του χρόνου ή σε δύο χρόνια με αφορμή αυτό το τραγικό δυστύχημα, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε περιπτώσεις ε, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον συντονισμό σε περιπτώσεις ε, ζήτησης ε, βοήθειας. Παραπάνω λεπτομέρειες δεν είμαι σε θέση να σας δώσω αυτή τη στιγμή, αλλά προσπάθησα να εκθέσω το γεγονότα με, την, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω που βρισκόμαστε ακριβώς, σε ποιο σημείο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω εγώ πρώτα πρώτα στο μυαλό μου. Ίσως εσείς κύριε Μίλη, μπορείτε να με ε, βοηθήσετε. Έχουμε όμως ένα πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο στο, στο πέλαγος και το μήνυμα το οποίο έχω λάβει είναι ότι όλοι ε, ένιψαν τα σχήρα του έκαναν τον πόντιο πιλάτο. Αυτό βέβαια, ό,τι κανονισμός και να υπάρχει, δεν λέει. Τα κράτη-μέλη, τα ίδια ένυψαν τα σχήρα τους. Είναι αλήθεια. Αν όμω είναι αλήθεια, τότε αυτή η αναθεώρηση, αυτή η μεταρρύθμιση, αν κατάλαβα καλά, τότε θα πρέπει αυτό ως ε, αλλαγή, ως μεταρρύθμιση στην νομοθεσία αύριο να, να, να, το προτείνετε. είναι δυνατόν να, έχουμε ένα κράτο μέλο το οποίο να, να λέει είμαι αρμόδιο ενώ ένα πλοίο κινδυνεύει. Το είχαμε ξαναυποστεί αυτό. Ε, κάποια στιγμή υπάρχει κάποιο κράτο μέλο το οποίο ακριβώ το έκανε το ίδιο πράγμα. Για το πλοίο που λεγόταν Prestige. Θυμάστε. Σα το λέω όσο πιο έντονα μπορώ. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο. Να μου το πείτε αν κάνω λάθο. Αλλά εάν έγινε κάτι τέτοιο, πλοίο το οποίο διατρέχει κίνδυνο ε, και ε, κράτη-μέλη ή, ή κράτος μέλος είπαν η τασίας μου δεν είμαι αρμόδιος, τότε αυτό είναι απαράδεκτο. Έχετε το λόγο κύριε Μίλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα συγχαρητήριά σας, ευχαριστώ για όλα όσα είπατε και πρώτα πρώτα θα πρέπει να σας αναφέρω ότι ορίστηκα, διορίστηκα στις 8 Ιουνίου στη θέση μου και μόλις πριν τρεις μέρες ανέλαβε τα μου, οπότε δεν έχω μπορέσει ακόμη να ενημερωθώ για όλα τα θέματα και δω τώρα ψάχνω περνασμένα στο, να συνδεθώ με τον υπολογιστή μου, να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία που τα έχει η ΕΜΣΑ για όλε αυτές τι αξιολόγες ερωτήσει και πρώτα πρώτα για την Φλαμίνια όπως είπε ο πρόεδρος, ε, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έγινε, μια που τα κράτη-μέλη να πετάνε τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Δεν ένα πλοίο, θα πρέπει αυτό το πλοίο να το πλησιώσει κανείς όσο γίνεται καλύτερα. Οπότε σε σχέση με αυτό, άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι πρέπει να το χέρι για να αναθεωρήσει τον κανονισμό και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μην έχουμε επανάληψη αυτού του θλιβερού φαινομένου. μπορεί να περιμένουμε περαιτέρω. Τώρα όσον αφορά την αυσιπλοεία αναφέρθηκε επανειλημμένα. Έχουμε κάποιους οι οποίοι ασχολούνται, κινούνται στον κλάδο αυτό και θα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε όλο ένα και νεότερους, περισσότερους να έρχονται στον κλάδο μας και ακριβώς όπως είπατε όχι μόνο στη γέφυρα αλλά και στο μηχανοστάσιο ό, όσο γίνεται περισσότερους γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε 75% τώρα ε, των, ε, των πληρωμάτων μας ε, που είναι από τρίτες χώρες. Άρα αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Γιατί βάλετε εκεί. κάτι είπατε και είπατε επίσης και για τον κόλπο της Φιλανδίας. Όντως, ευαίσθητη περιοχή συνολικά. Θα τριπλασιαστεί η κίνηση, μια που οι Ρώσοι στο νότιο του κόλπου της Φιλανδίας... Ε, θα έχουν το Σλούγκα με ένα νέο λιμάνι που θα διακινεί πάρα πολύ μεγάλα φορτία. Και έτσι έχουμε 100 εκατομμύρια τόνους φορτίου μόνο εκεί. Επομένως γι' αυτό και είναι πάρα πολύ βασικό μας θέμα η, η ασφάλεια, το να μπορούμε να ολοκληρούμε και ναι, να μπορούμε να, να, να κινούμεθα στις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες αυτών των περιοχών η Εστονία, Ρωσία και οι άλλες χώρες που βρέχονται από αυτά τα νερά έχουν προσπαθήσει σε συνεργασία να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και πώς θα, θα είναι δυνατόν να βελτιωθεί η, η ασφάλεια. Και βέβαια, πάντοτε έτσι υπάρχει ε, ο κίνδυνος του να σπεύσει κανείς βραδέως, γιατί όπως με τα πράγματα, η καλύτερη προστασία είναι εκ των προτέρων και από την ξηρά κανείς να το φροντίσει. Και να δούμε το πόσον εδώ το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, και για την ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε τι γίνεται με τη στρατηγική τη Βαλτική θάλασσα. Και βέβαια η ασφάλεια της ναυσιπλοείας ασφαλή στη θάλασσα είναι ο πυλώνας της πολιτικής αυτής. Επίσης, μεγάλη μου χαρά, άκουσα τα όσα είπατε υπέρ του έργου μας και στο μέλλον θέλουμε να έχουμε στενή συνεργασία με το Κοινοβουλίο συγκεκριμένα με την Επιτροπή σας και με όλες τις, ε, ε, τις επιτροπές, όλα τα, τα θεσμικά όργανα. Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας αυτή θα οδηγήσει στην επιτυχία του έργου μας. το τι γίνεται με τα κράτη-μέλη. Το 2012 Είχαμε έξι δράσεις κατάρτισης, 270 επομένως ε, αξιωματικοί, αξιωματούχοι ε, παραγούσαν την ε, εκπαίδευση και εμείς θα συνεχίσουμε για αυτόν τον τρόπο. παρακολουθούμε τι γίνεται στα κρατημέλη. Και έτσι ελπίζουμε στο μέλλον να κάνουμε το μικρό. Τη Φλαμίνια. Για άλλη μια δουλειά, για άλλη μια φορά να σας αναφέρουμε ότι δεν μπορούμε να παρεμβούμε. Είναι θέμα κρατών μελών. Γιατί είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό αφορά και τη διάσωση πλέον. Πάντως, που είναι κατάπληξη αυτό το οποίο έγινε. Είναι απαράδεκτο. 100% όπως τα είπε ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Ε, είπατε για αυτή τη θητεία θα είναι συνολικά δεκαετής. Εμείς πάντως θα είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί σας για ανταλλαγή πληροφοριών και βεβαίως θα δεχθούμε την ευγενή σας πρόταση. Θα έρθει μια μικρή μας αντιπροσωπεία να σας επισκεφθεί. Ναι, το πρόβλημά μας είναι πάντως η ατζέντα μου που έχει τόσο, τόσο, τόσο πολλές υποχρεώσεις που ματιώνει κάθε τέτοια προσπάθεια. Πάντως έτσι κι αλλιώς σας ευχαριστούμε που ήρθατε και απομαντήσατε και τις ερωτήσεις μας διευκρινίσατε τι ισχύει για το Φλαμίνιο Μάλιστα. συντονιστέ, τώρα, ε, σας δίνουμε λοιπόν πέντε λεπτά για να αδειάσετε την αίθουσα και έπειτα θα συνεχίσουμε με τι συνεδρία των συντονιστών.